Ja, Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ας προσέλθει και ο γερμανο γερμανο-ισπανικός συνασπισμό που μόλις μπαίνει στην αίθουσα. Να αρχίσουμε εδώ τη δεύτερη, το δεύτερο μέρος της ε, σημερινή συνεδρίας μετά από την ψηφοφορία που μάλιστα είχε και ενδιαφέρουσες πλειοψηφίες και ερχόμαστε τώρα στα θέματα Ρουμανία-Βουλγαρία και ελεύθερη, διακίνηση των εργαζομένων. Το ιστορικό είναι σαφές. Έχουμε στη διάθεσή μας μια δυναμική αγορά εργασίας, αλλά με πολλούς φραγμούς από πλευράς χωρών μελών και στις χώρες μέλη δηλαδή. Όσοι λοιπόν τα δραστήρια άτομα, 9 από 27 χώρες μέλη δεν έχουν ακόμη ελευθερώσει την διακίνηση των Ρουμάνων και Βουλγάρων επικών. Είναι σωστό αυτό, πρέπει να παρεμποδίζει τη κινητικότητα ορισμένων πολιτών. Η σημαντική ανεργία σε αριθμό, δηλαδή περίπου 10% κατά μέσον όρο, θα ε, μειωθεί με τον τρόπο αυτό. Εμίνιον Ντασίλβα ήθελε να έλθει, όπως μας ειδοποίησε, αλλά βρίσκεται στη Δανία, στο Συμβούλιο ΕΠΣΟ. Έχουμε όμως τον τμήματάρχη του, της Κομισιόν για την πρώτη τοποθέτηση για να μπορέσουμε στη βάση αυτή να προχωρήσουμε σε μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα πολύ γρήγορα να σας παρουσιάσω μερικές πληροφορίες σε σχέση με την κατάσταση αυτού του φακέλου. Ζητώ συγγνώμη για την απουσία του κυρίου Σίλβα. Υπενθυμίσατε κι εσείς, έχουμε μεταβατικά μέτρα για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, τα οποία εισήχθηκαν κατά την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας το 2007 μέτρα μέγιστης διάρκειας 7 ετών, τα οποία περιλαμβάνουν τρεις φάσεις. Η τελευταία φάση, η διάρκεια 2 ετών, ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο. Η εισαγωγή μεταβατικών μέτρων δεν αφορά συγκεκριμένα αυτή την τελευταία διεύρυνση. Και στις παλαιότερες διευρύνσεις ε, εισήχθησαν παρόμοια μέτρα, τα οποία αποσκοπούσαν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για αυτή τη διεύρυνση. Η εισαγωγή τέτοιων μέτρων ε, είναι ωστόσο ανευαίσθητο θέμα διότι αφορά την άσκηση μιας θεμελιώδους ελευθερίας, της ελευθερίας ε, ε, κυκλοφορίας των εργαζομένων. Όσον αφορά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η τρίτη φάση των μεταβατικών μέτρων που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2012 θα ολοκληρωθεί αμετάκλητα στις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Πριν από εκείνη την ημερομηνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο εκθέσεις για τη λειτουργία αυτών των μεταβατικών μέτρων. Η πρώτη συμμορφωνόταν με τη συνθήκη ένταξης ήδη τον Νοέμβριο του 2008 και μια δεύτερη έκθεση τον Νοέμβριο του 2011 μετά από αίτημα των δύο ενδιαφερομένων χωρών. Η εν λόγω έκθεση εγκρίθηκε από την Κομισιόν τον Νοέμβριο του 2011. Έστελνε μια σειρά μηνυμάτων, ειδικότερα το γεγονός ότι η κινητικότητα από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία επηρεάζει θετικά από οικονομική άποψη τόσο την αύξηση όσο και τις δυνατότητες ε, κάλυψης ε, ελλείψεων ε, εργαζομένων στα κράτη-μέλη ότι έχει περιορισμένες επιπτώσεις στους μισθούς και στην απασχόληση των εργαζομένων στις χώρες υποδοχής ότι η μείωση της αίτησης της ζήτησης εργαζομένων μείωσε τη ροή εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και ότι η υλοποίηση των μεταβατικών μέτρων επηρέασε σε μικρό βαθμό την κινητικότητα, τις ροές κινητικότητας. Η κινητικότητα αυτή επηρεάζεται ουσιαστικά περισσότερο από άλλους παράγοντες όπως οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας, η ύπαρξη δικτύων υποδοχής ή η γλώσσα. Οι συνθήκε ένταξη τη Βουλγαρία και τη Ρουμανίας προβλέπουν ότι τα κράτη-μέλη που έχουν διατηρήσει περιορισμού στη δεύτερη φάση μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτού του περιορισμού και κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης, δηλαδή από τον Ιανουάριο 2012 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013, σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων ή σοβαρών κινδύνων ε, ύπαρξης προβλημάτων στην αγορά εργασίας τους. Σε τέτοια περίπτωση ήταν υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν ε, την Κομισιόν για την πρόθεσή τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν υπήρχε για τα 11 κράτη-μέλη που είχαν συνεχίσει μέχρι τα τέλη του 2011 να εφαρμόζουν αυτές τις εθνικές συνθήκες για την πρόσβαση στην αγορά εργασία τους, αγορά εργασίας τους για τους Βούλγαρους και Ρουμάνους εργαζομένους. Στα 11 αυτά κράτη-μέλη, δύο η Ιταλία και η Τσεχική Δημοκρατία ενημέρωσαν για την απόφασή τους να εφαρμόσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στους Βούλγαρους και Ρουμάνους εργαζομένους ε, από τον 1η Ιανουαρίου του 2012. Τα άλλα 11 κράτη-μέλη, ε, τα άλλα 9 κράτη-μέλη, συγγνώμη, η Γερμανία, Η Ιρλανδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, κάτω χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Μάλτα και Αυστρία, έστειλαν ειδοποίηση στην Κομισιόν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 για να ενημερώσουν ότι έχουν λάβει απόφαση να συνεχίσουν την εφαρμογή των εθνικών μέτρων και εξηγώντα ε, ότι αντιμετωπίζουν ε, αναταραχές προβλήματα στην αγορά εργασίας τους ή κινδύνους σοβαρών προβλήματων στην αγορά εργασίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησε προσεκτικά τις ε, ειδοποίησεις αυτές που έλαβε τόσο από τις τυπικές πτυχές όσο και για το περιεχόμενό τους. Όσον αφορά τις ε, τυπικές πτυχές, ε, τα εννέα κράτη-μέλη τήρησαν όλα τις προθεσμίες και συνόδευσαν τις ε, ειδοποιήσεις τους με επεξηγηματικά στοιχεία για τους λόγους που επιβάλλουν τους περιορισμούς και ποσοτικά μεγέθη που σχετίζονται με την κατάσταση της αγοράς εργασίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε το περιεχόμενο αυτών των εκθέσεων εξέτασε τη συνοχή των δικαιολογητικών και την ποιότητα των πληροφοριών που τις υποστηρίζουν. Τα κυριότερα επιχειρήματα που παρουσίασαν τα κράτη-μέλη αφορούσαν την τρέχουσα κατάσταση και τις δυσίωνες προοπτικές των οικονομιών και των αγορών εργασίας στα ενδιαφερόμενα κράτη κράτη-μέλη, ειδικότερα όσον αφορά την ανάπτυξη, το ποσοστό ανεργίας, την αρνητική εξέλιξη των προσφορών θέσεων εργασίας. Ένα δεύτερο επιχείρημα αφορούσε τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με το άνοιγμα της αγοράς εργασίας σε ορισμένους τομείς, σε ορισμένες ομάδες εργαζομένων ή σε ορισμένες περιφέρειες. Ειδικότερα υπογραμμίστηκαν οι κίνδυνοι αυτού του ανοίγματο για τους ήδη εγκατεστημένους μετανάστες σε αυτά τα κράτη που επηρεάζονται περισσότερο από τους υπόλοιπους, από την ανεργία και ενδεχομένως έρχονται σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό με τους ε, παρομοίως ε, αναφερόταν ε, το υψηλό ποσοστό, ο κίνδυνος υψηλό ποσοστό ενεργείας. Ε, τα εννέα κράτη-μέλη υπογράμμισαν επίσης τον κίνδυνο διαφοροποίησης των ροών κινητικότητας σε περίπτωση ε, ανοίγματο που δεν ακολουθηθεί από άλλες χώρες. Ειδικότερα η απόφαση της Ισπανίας να ενεργοποιήσει τη ρήτρα ε, διασφάλισης τον Ιούλιο του 2011 και η αβεβαιότητα για τι αποφάσει των γειτονικών κρατών σίγουρα επηρέασαν τι αποφάσει ορισμένων κρατών μελών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία και το Λουξεμβούργο, αποφάσισαν να αλαφρύνουν τους περιορισμούς και να ανοίξουν περισσότερο τις αγορές εργασίας τους. και ενημέρωσαν για αυτό ε, στο παράρτημα που συνόδευε την ειδοποίηση που απέστειλαν. Από καθαρά τυπική άποψη η παράταση των μεταβατικών μέτρων στην τελευταία φάση δεν απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα κράτο μέλο το οποίο ειδοποιεί εντό προθεσμία την απόφασή του να συνεχίσει την εφαρμογή των μεταβατικών μέτρων δεν χρειάζεται καμία άλλη έγκριση. Η Κομισιόν είχε ωστόσο ειδοποιήσει τα κράτη-μέλη τον περασμένο Νοέμβριο για την ανάγκη ε, επισύναψης πολύ λεπτομερών επιχειρημάτων προς υποστήριξη των ειδοποιήσεων. Κατά την, ε, σε βάθος μελέτη, περίπτωση κατά περίπτωση αυτών των ειδοποιήσεων, η Κομισιόν εκτίμησε ότι τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη παρουσίασαν επιχειρήματα με συνοχή και που συμμορφώνονται με τους νόμους. Στις 17 του περασμένου Φεβρουαρίου παρουσιάστηκαν ε, οι αποφάσεις στο Συμβούλιο, σημειώθηκαν οι αποφάσεις και τα επιχειρήματα των κρατών μέλων και η συμμόρφωση των ειδοποιήσεων αυτών. Ωστόσο, ε, θεώρησε ε, σκόπιμο να μεταδώσει τα εξή μηνύματα, μεταξύ των οποίων αυτό που σχετίζεται με το γεγονό ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή, ότι είναι υποφελής τόσο για τους εργαζομένους όσο και για το σύνολο τη οικονομία. Το γεγονός επίσης ότι δεν έχει αποδειχθεί πως το άνοιγμα των συνόρων για τους κοινοτικούς εργαζομένους αποτελεί αρνητικό ε, στοιχείο για την αγορά εργασίας και το γεγονός επίσης ότι οι ροές κινητικότητας τροφοδοτούνται κυρίως από τη ζήτηση εργαζομένων και ότι η κινητικότητα είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός κάλυψης των ελλείψεων εργατικού δυναμικού. Αυτή η πτυχή επίσης υπογραμμίστηκε σε μια ανακοίνωση της Κομισιόν της 18 Απριλίου για τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση, όπου γίνεται έκκληση προς τα κράτη-μέλη για άρση των περιορισμών. Τέλος, ο επίτροπο επίσης υπογράμισε ότι ο περιορισμός τη ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες, ειδικότερα σε εποχέ κρίσης, διότι μπορεί να επηρεάσει τις ε, συμπεριφορές, αμφότερες συμπεριφορές και να ενθαρρύνει την παράνομη εργασία. Μετά από αυτό το Συμβούλιο, ο Επίτροπος Αντόρ έστειλε τα σχόλιά του εγγράφου στα εννέα κράτη-μέλη, στα εννέα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, στα μέσα Μαρτίου. Στην επιστολή του υπενθύμησε εκτός των γενικών σχολείων το νόημα των μεταβατικών μέτρων που είναι να δίνουν στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να προετοιμάζονται βαθμιαία για το πλήρες άνοιγμα των συνόρων και όχι να καθυστερούν ε, και να τηρούν τις προθεσμίες μέχρι το τέλος. Υπενθύμησε λοιπόν στα κρατη έκανε έκκληση προς τα κράτη-μέλη να επαναξιολογούν διαρκώς τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας τους και να επανεξετάζουν συνεχώς το κατά πόσο αρμόζει να διατηρούν τις ε, περιορισμούς και κατά πόσο θα πρέπει να τους αλαφρύνουν κατά τις τελευταίες φάσεις ε, έως τα τέλη του 2013. Επίσης ε, κάλεσε μια σειρά κρατών μελών να συμπληρώσουν από εδώ, από τώρα μέχρι τα μέσα Μαΐου, μια έκθεση προς την Κομισιόν προσφέροντας περισσότερες προφορές για την αγορά εργασίας, ώστε να υποστηρίξουν ε, την επιχειρηματολογία τους όσον αφορά τα προβλήματα στις αγορές εργασίας. Τέλος, ο Επίτροπος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ε, υπάρξει μία μελέτη σε ενδιάμεση φάση, στη μέση περίπου της εφαρμογής των ε, μεταβατικών μέτρων. Η Κομισιόν λοιπόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα εννέα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη έως τα τέλη του 2013. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε της Κομισιόν. Αρχικά είχαμε σχεδιάσει μέχρι παρατέταρτο, δηλαδή 20, λεπτά ακόμη να... Α, βλέπω και τον κύριο Κώσα που ζητεί το λόγο. Θα σας πω τώρα τα ονόματα που έχω εγγράψει είναι τα εξής. Αυτά είναι τα πρόσωπα που ήδη ζήτησαν το λόγο και έχουν εγγραφεί. από τη Ρουμανία, η κυρία Πλάμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω ρουμανικά. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μήνυμα που μας διαβίβασε από τον ε, Επιτροπό του κύριο Άντορ την επισκόπηση δηλαδή της καταστάσεως σχετικά με τους περιορισμούς από πλευράς αγοράς εργασίας για εργαζόμενους Ρουμάνους και Βουλγάρους. Εγώ έχω το εξή μήνυμα και θα ήθελα επίσης να απευθύνω και μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα, βέβαια, μιλούμε, αναφερόμαστε εδώ δηλαδή, στις αρχές που αποτελούν το θεμέλιο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ελευθερία διακίνησης των εργαζομένων. Εγώ θα ήθελα ωστόσο να μιλήσω για την κινητικότητα πρώτα-πρώτα των εργαζομένων που θεωρώ ότι αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει απασχόληση, μπορεί να σταθεροποιήσει την αγορά εργασίας. Εγώ νομίζω ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις που να επιτρέψουν οι όροι που επιβάλλονται στις αγορές, σύμφωνα δηλαδή με τις συνθήκες εντάξεις Βουλγαρίας και Ρουμανίας, και μιλώ για τα μεταβατικά μέτρα βεβαίως, οι όροι αυτοί λοιπόν που εν τέλει προκαλούν διακρίσεις και που μόνο αρνητικά αποτελέσματα έχουν, αρνητικές επιπτώσεις έχουν και στην αγορά εργασίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα, αυτοί οι όροι πρέπει να καταργηθούν. Πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί για τους Ρουμάνους και Βουλγάρους εργαζομένους. Για μας είναι πολύ σημαντικό, ιδίως σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου καλούμαστε να αναζητήσουμε τις καλύτερες λύσεις για να μπορέσει η Ευρώπη να βγει από την κρίση, πρέπει να εξασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης κατάλληλες που να προσφέρουν αξιοπρεπή εργασία και συνθήκες διαβίωσης. Και όχι να διατηρούμε εξαιρέσεις. Μας έδωσε την απάντηση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ότι ένα από τα επιχειρήματα που επικαλούνται λέει ότι με την κινητικότητα Βουλγάρων και Ρουμάνων στην αγορά εργασίας μπορεί να προκληθούν ανισορροπίες. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να εξαλειφθεί. Πρέπει να βρούμε βιώσιμες λύσεις να δούμε δηλαδή ποιε είναι πρώτα-πρώτα οι αληθινέ αιτίε τη κρίση, όπω γνωρίζουμε όλοι, οι αληθινέ αιτίε τη Κρίση δεν έχουν καμία σχέση με το άνοιγμα των αγορών εργασία στου Ρωμάνου και Βουλγάρους. Είναι σαφή, λοιπόν η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Με την κινητικότητα των εργαζομένων θα υπάρξουν ευεργετικά αποτελέσματα, μάλλον, και όχι το αντίθετο. Γι' αυτό και θέτω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από, την, από τις απαντήσεις που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα Μαΐου, θα διεξαχθεί νέα αξιολόγηση. Θα δοθεί συνέχεια στα επιχειρήματα αυτά. Θα επανεξετάσουν την απόφαση που έχει σχέση με την κινητικότητα των εργαζομένων από Ρουμανία και Βουλγαρία. Ευχαριστώ κυρία Πλάμ. Μία συνάδελφος, η κυρία Στάινρουκ. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ σε όλα όσα είπε η κυρία Ροβάνα Πλάμ. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Γερμανία είναι μία από τις χώρες εκείνες η, οποία ε, επιβάλλει ακόμα σημαντικούς περιορισμού στην διακίνηση εργαζομένων από η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Αυτό αντιβαίνει στην ελευθερία διακίνηση των εργαζομένων, σύμφωνα με την άποψή μου και την άποψη της πολιτικής μου ομάδας των σοσιαλδημοκρατών. Η θέση μου και η θέση του γερμανικού S5 είναι ότι τα προβλήματα δεν προκαλούνται από την ελευθερία διακίνησης. Στη Γερμανία είναι περισσότερο οι αιτίες η έλλειψη κατώτατου μισθού, η διάφοροι τρόποι με τους οποίους προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα οι ψεύδο ανεξάρτητοι επαγγελματίε και άλλα σχετικά θέματα. Τώρα, εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτα, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δηλώνει ότι φοβάται ότι θα εκτοπιστούν από την αγορά εργασίας εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι, προσοντούχοι εργαζόμενοι, όταν θα προσέλθουν οι εργαζόμενοι από τις χώρες αυτές. Επιβεβαιώνεται η εμπειρία αυτή από την εμπειρία άλλων, ο φόβος αυτός, συγγνώμη, από την εμπειρία άλλων χωρών. Το άλλο είναι, το άλλο επιχείρημα είναι, της γερμανικής κυβέρνησης, ότι θέλει να αποφύγει το dumping στο, στους μισθούς και στις κοινωνικές εισφορές. Πάλι εδώ ερωτώ, ποιες είναι οι εμπειρίες άλλων χωρών μελών που έχουν επιτρέψει την ελεύθερη διακίνηση και ιδίως σε ό,τι αφορά και τους κατώτατους μισθούς. Ευχαριστώ, Γιούτα. Ο κύριος Κλάρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι ο μόνος που παρατηρεί ότι η διευθέτηση μεταβατική εκπνέει το 2013 και θα έλεγα ότι και μία από τις βασικές εφημερίδες της χώρας μου το έθεσε με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ανοίξει τις πύλες του Ηνωμένου Βασιλείου να εισρεύσουν εργαζόμενοι». Φοβούμαι ότι γινόμαστε, γινόμαστε στόχος και ε, τα ποσοστά ανεργίας αυτή τη στιγμή είναι στο 8,3%. Στη Βουλγαρία 12%. Οπότε βλέπω το κίνητρο για αυτή τη μετακίνηση. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι πολύ περισσότεροι Ρουμάνοι και Βουλγαροί πηγαίνουν σε Ισπανία και Ιταλία παρά στην Ουκρανία. Όμω Ιταλία και η Ισπανία αυτή τη στιγμή σφυρο από την οικονομική κρίση. Η Ισπανία έχει ξεπεράσει 40% τη ενεργεία μεταξύ των νέων. Βλέπω λοιπόν άνθρωποι από την Ανατολική Ευρώπη καλό να το ξανασκεφτούν και να επιλέξουν χώρες με καλύτερε προοπτικέ σε ό,τι αφορά την απασχολησιμότητα, όπως εμείς. Δεν μου φαίνεται λοιπόν περίεργο όταν ε, γίνονται εχθρικοί οι συμπολίτε μου ένα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προηγούμενη χρονιά, ε, μια έκθεση έλεγε ότι οι Βρετανοί εργαζόμενοι έχασαν 166.000 θέσει εργασία. Ταυτόχρονα κερδίθηκαν 166.000 θέσει εργασία από αλλοδαπού είναι σύμπτωση αυτή η ταύτη αριθμών, όμω δείχνει μία τάση. Και πριν σχηματίσετε λανθασμένη εικόνα για μένα και τη θέση μου, να εξηγήσω το εξή. Εμείς έχουμε δεχτεί άλλους ανθρώπους από όλα τα μέλη του κόσμου εδώ και αιώνες, αλλά σε σχετικά μικρούς αριθμούς ώστε να μπορούν να αφομοιωθούν, να γίνουν κομμάτι της κοινωνίας μας, να γίνουν εμείς οι ίδιοι, να γίνουν η κοινωνία που είμαστε σήμερα, καθώς αυτές οι εισφορέ έγιναν βαθμία και μικρός αριθμό. ενώ αντίθετα σήμερα βλέπουμε 200.000 ετησίω. Όταν κανεί ερχόταν πριν από δύο αιώνε, δεν χρειαζόταν περισσότερε υπηρεσίε, γιατρού, ε, εκπαίδευση, δρόμου κτλ. Γιατί αρκούσαν ήδη. Όμω σήμερα χρειάζομαστε πιο πολλέ υπηρεσίε. Πού θα τι βρούμε, σήμερα στη πιο πυκνοκατοικημένη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόνο αυτό δείχνει πώς είναι μη βιώσιμη κατάσταση. Παρακαλώ και πάλι μη σχηματίστε λανθασμένη εικόνα από αυτά που λέω. Να σας δώσω μια προσωπική μου άποψη. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Έχω διδάξει εδώ και 39 χρόνια. Συνταξιοδοτήθηκα το 1983 και όταν συνταξιοδοτήθηκα κοίταξα πίσω την καριέρα μου και συνειδητοποίησα το εξής με την πιθανή εξαίρεση της Λατινικής Αμερικής, δίδαξα παιδιά από όλο τον κόσμο. Όμως είναι τα παιδιά οικογενειών από όλο τον κόσμο. Από την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ινδία, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Καναδά, Αμερική, ε, Δυτικές Ινδίες, Αφρική και ναι, από την Ευρώπη, την Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Νορβηγία, Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία. Ήταν όλοι ευπρόσεκτοι στα σχόλια μας. Ήταν χαρά να διδάσκει σε αυτά τα παιδιά. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι να δεχτούμε αυτούς τους αριθμούς που βλέπουμε σήμερα. Και κλείνοντα να κάνω ένα σχόλιο, μου επιτρέπετε, Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει ρητά ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κανενός είδους στην Επιτροπή μας μόλις σήμερα το πρωί, στην έκθεση ΧΙΕΣ, είδαμε με μια προφορική τροπολογία της εισηγήτριας που έτυχε ευρεία στήριξη και υιοθετήθηκε, που έλεγε ότι θα είναι μηδενική η ανοχή στι διακρίσει, στην κρατική μεταχείριση. Και όμω, τι βλέπει κανεί αυτή την έκθεση τη Κομισιόν που συζητούμε αυτή τη στιγμή, στην παράγραφο 1-3, πρώτη σελίδα ένα κράτος μέλος πρέπει πάντοτε να δίνει προτίμηση σε Βουλγάρους και Ρουμάνους εργαζόμενους έναντι, με, ε, ε, μάλλον έναντι υπηκών ε, μη ευρωπαϊκών χωρών. Άρα δηλαδή εμείς θα πρέπει να κλείσουμε τις πόρτες από τους φίλους από την κοινοπολιτεία. Αυτό δεν είναι διακριτική μεταχείριση, πρόεδρε. Ελπίζω να είστε περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Κλάρκ. Κύριε Κορνέλησεν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, συγκινητική αυτή η ιστορία, από την οποία θα επιλέξω τις ε, ε, χαρούμενες θυμίσεις της διδασκαλίας σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο και τα υπόλοιπα δεν ε, θέλω να τα διατηρήσω στο μυαλό μου. Χαίρομαι πολύ για την επιστολή που εστάλει ο κύριο Αντόρ το είχε υποσχεθεί στα τέλη του περασμένου έτους και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που έχει σταλεί. Θα ήθελα να δω ένα αντίτυπο αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε ποιες ε, ε, χώρες, σε ποιες χώρες, ποιες χώρες ζήτησαν, ε, σε ποιες χώρες ζητήθηκε περισσότερη απόδειξη για τα προβλήματα στις αγορές τους. Έχουν ληφθεί απαντήσεις και ποια είναι η προθεσμία. Τόσο, όσον αφορά το περιεχόμενο θα ήθελα να μου πείτε τι συνιστά καλό επιχείρημα διότι βάσει πολλών ερευνών λέγεται ότι οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι δεν δημιουργούν προβλήματα διατραχές στις αγορές εργασίας και ειδικότερα όχι σε χώρες που πάνε ιδιαίτερα καλά όπως οι χώρες και η Γερμανία. Δεν καταλαβαίνω πού θα μπορούσαν να βρουν επαρκή επιχειρήματα για να αποδείξουν κάτι τέτοιο. Η δεύτερη ερώτηση, χαίρομαι ιδιαίτερα που θα υπάρξει μια ενδιάμεση έκθεση Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, δείξουμε πως ε, ε, όταν επηρεάζουμε ένα σημείο τα αποτελέσματα φαίνονται κάπου αλλού στις κατοχώρες έχουμε ήδη δει ότι τα περιοριστικά μέτρα έχουν οδηγήσει σε 16% 16% περισσότερου αποσπασμένου και αρκετό μεγάλο ποσοστό περισσότερων ε, ελεύθερων επαγγελματιών μεταξύ Βουλγαρών και Ρουμανιών και ξέρω ότι ένα μεγάλο ποσοστό ε, Ρουμάνων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτεπάγγελτοι το οποίο είναι εξωφρενικά υψηλό ποσοστό σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλε χώρες. Θα ήθελα να πείτε ε, λοιπόν κατά πόσο μετά από παρακολούθηση θα προκύψουν τα ίδια ποσά. Και το τελικό ερώτημα είναι τι θα γίνει στη συνέχεια. Για να σας πω για τις κατοχώρες, είδα την επιστολή που έστειλαν για την ειδοποίηση. Ήταν αρκετά αστεία. Στο τέλος αναφερόταν ότι σχεδόν κανένας Βούλγαρος και Ρουμάνος δεν χρησιμοποιεί την κοινωνική ασφάλιση στις κατοχώρες, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει. Αυτό αποτελεί επιχείρημα. Είμαι αρκετά βέβαιη ότι θα πρέπει κάποιο να του έστειλε μια επιστολή ζητώντα περισσότερε εξηγήσει και είμαι βέβαιη ότι θα απαντήσουν ε, χωρί να έχουν περισσότερα επιχειρήματα. Και τι θα γίνει μετά στη συνέχεια. Ε, Σα ευχαριστώ, Μαρία. Ο κύριο Κώστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μου δίνετε το λόγο. Αυτή τη στιγμή παίρνω το λόγο εξ ονόματος ε, του συντονιστή του ΕΛΚ, του κυρίου Όρη, ο οποίος ε, δυστυχώς δεν μπορεί να σήμερα παρόν. Είμαι της γνώμης ότι οι προλαλήσαντες ε, έθεσαν πολύ σημαντικά επιχειρήματα για το θέμα που ζητούμε αυτή τη στιγμή. Κατά μένα τα πράγματα είναι σαφή. Μιλάμε για μια βασική αρχή που διέπει ε, τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο περιορισμός ε, στην εφαρμογή μιας τέτοιας αρχής θα πρέπει να δικαιολογείται παρκώς και οι εξηγήσει τώρα είναι επαρκή. Το 2006 ε, ασχολήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το θέμα αυτό και επισημάνθηκε ότι τέτοιου είδους περιορισμοί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους στόχους για τους οποίους ε, ευθύς εξ αρχής ε, αποφασίστηκαν. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αναλυθούν δράσεις και όχι να γίνουν αυτοί περιορισμοί. Αντίθετα, πρέπει να ληφθούν δράσεις προ όφελο των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη, για να δημιουργηθούν θέσει εργασία, να έχουμε κινητικό των εργαζομένων και να υπάρχει ισορροπία. Αυτή είναι η στόχη που πρέπει να επιτύχουμε. Χαιρετίζουμε τα βήματα που έκανε ως τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε της γνώμης ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. ώστε να μπορούν να αρθούν πλήρως οι περιορισμοί αν είναι δυνατόν και νωρίτερα από το 2013. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Ο κύριο Σέρκας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ μιλώ εξ ονόματός μου, αλλά και εξ ονόματος πολλών συναδέλφων ε, της ομάδας ε, των σοσιαλιστών. Πρώτα απ' όλα μια προσωπική σκέψη θα ξεκινήσω, που θεωρώ ότι έχει μια βάση από μακρά ε, χρονική εμπειρία. Πλησιάζει αυτή η ημερομηνία της φάσης μεταβατικής περίοδου και θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι αυτή η συζήτηση είναι μοναδική τροποντινά. Σε αυτή την Επιτροπή συχνά μιλάμε για τη δικαιώματα των εργαζομένων. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά για μία από τις θεμελιώδες από τις ελευθερίες ελευθερίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παράδοξο τροποντινά θα έλεγα και καταλήγει να σοκάρει θερός ότι είναι σκανδαλώδες κατά με ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλάμε και να περασπιζόμαστε τις οικονομικές ελευθερίες και να τις βάζουμε πάνω από τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και μάλιστα τώρα αυτές αυτά τα δικαιώματα να τα βάζουμε και πάνω από τα θεμελιώδη δικαιώματα, θεμελιώδες ελευθερίες. Και έτσι να δίνουν μια πολύ αρνητική χρειά σε αυτή τη βασική αρχή που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να τα πούμε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κλαμπ όπου όλοι μπήκαμε θελοντικά. Όποιο λοιπόν έχει μπει μέσα θα πρέπει να τηρεί του κανόνε αυτό το κλαμπ. Αλλιώ να σηκωθεί να φύγει. Αν παραμένει μέσα θα πρέπει να τηρεί του κανόνε που ισχύουν εδώ υπερασπιζόμαστε τις ελευθερίες γενικότερα, ναι, αλλά υπερασπιζόμαστε την ελευθερία να ανοίγει κανείς ένα κατάστημα που σερβίρει ουίσκι, ε, ένα σούπερ μάρκετ κτλ. Ωραίες όλες τις ελευθερίες, αλλά από την άλλη υπάρχουν και τα δικαιώματα των εργαζομένων και προκειμένου μιλάμε για ελευθερίες, μιλήσω ελευθερίες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια εξαίρεση, όπω είπε και πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου, επταετία για την προετοιμασία των κρατών μελών και για να μπορέσουν να φτάσουν σε μια χρονική στιγμή, πλέον μετά από αυτήν την εφταετία, ώστε να μην ακούμε έτσι ανενδίαστα και ξεδιάντροπα τέτοιου είδου θέσει. Ποιο μιλάει για χιονοστιβάδα εργαζομένων από αυτέ τι χώρε, όταν υπάρχουν χώρε που άνοιξαν νωρίτερα τα σύνορά του και δεν πλημμυρίστηκαν από κανέναν. Όταν έχουμε 350 εκατομμύρια ε, ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, εργαζομένους από αυτές τις δύο χώρες αν ο επιμερισμός και η κατανομή γίνει ισότιμα το πρόβλημα υπάρχει. Γι' αυτό και εμείς προβήκαμε στη θέσπιση ενός συντηρητικού μέτρου. Αν κλείσουν τα σύνορα κάποιοι, τότε θα δούμε ανισορροπίες. Αν όμως ο καθένας είναι διαθέσιμος να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης του και να δεχθεί εργαζόμενους που θα έρθουν να βοηθήσουν στις οικονομίες μας, δεν θα μας πλημμυρίσει και θα μας πείσει κανένας. Και κάτι άλλο που θεωρώ τον δραματικό πρόεδρε και το ακούμε δυστυχώς σήμερα, από το στόμα της ακροδεξιάς, από τη γαλλική προεκλογική στρατεία είναι ότι αυτοί θα πρέπει να φύγουν οι εργαζόμενοι για να αφήσουν τη δουλειά στους ε, ντόπιου εργαζόμενους. Μα αυτοί οι άνθρωποι κάνουν δουλειές που δεν επιθυμούν να κάνουν οι μεδαποί. Να μαζεύουν τα σκουπίδια, να φροντίζουν ηλικιωμένους και άρρωστους κτλ. Πρόκειται για εργασίες που δεν επιθυμούν να κάνουν ε, οι μεδαποί. Και θεωρώ ότι τέτοιου είδους απόψεις προκαλούν ντροπή. Είναι ντροπή και δεν ευσταθούν σε καμία περίπτωση για τους θέσεις. Και τέλος, πρόεδρε, θεωρώ ότι έναντι αυτών των σοκαριστικών δηλώσεων, θέλω να πω, και εμεί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ απίφθηνα μια έκκληση στον Επίτροπο Άντρο και απευθύνω μια νέα έκκληση. Τα νέα κράτη-μέλη που ανακοινώνουν ότι θα συνεχίσουν α, να εφαρμόζουν τα περιοριστικά μέτρα και το 2014, να πούν στην Κομισιόν κατά πόσον έχουν συνεκτικά και ακόλουθα στοιχεία για το αυτό. Όταν στην επιστολή Επιτροπή λέει ότι δεν έχουν υποστεί αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας τους έως σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι όταν η αγορά εργασία πάσχει σε μια χώρα, ε, δεν πηγαίνουν σε αυτή τη χώρα είναι οι εργαζόμενοι. Στη χώρα μου υπάρχει έλλειψη προσφορά θέσεων εργασία. Ε, λοιπόν, οι μετανάστε σηκώνονται και φεύγουν. Όταν δεν υπάρχει εργασία, δεν υπάρχει επιπρόσθετο πρόβλημα. Αυτό που θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εξή και το λέω εξ ονόματο ε, τη Σοσιαλιστική Ομάδα ότι θα πρέπει να είστε πιο κατηγορηματικοί στη θέση σα. Γιατί εσεί είστε ο θεματοφύλακα των συνθήκων, μιλάμε για μια θεμελιώδη ελευθερία και δεν υπάρχει κανένα ισχυρό στο επιχείρημα πέρα από τις προκαταλήψεις και τις ιδιοληψίες, ε, τις ακραίες ιδιοληψίες. Κανένα σοβαρό επιχείρημα που να στέκει ώστε μετά από 7 χρόνια να μην έχει τα σύνορα της Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην λέει ότι υπάρχουν ακόλουθα στοιχεία όταν όλα είναι ανακόλουθα ε, σε αυτόν τον ισχυρισμό. Ευχαριστώ κύριε Σέρκας. Η κυρία Ζίπελ, προτελευταία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με προκάλεσαν ορισμένε από τις δηλώσεις που άκουσα να επανέλθω. Και μετά τα όσα είπε ο κύριος Σέρκας, εγώ θα πω ότι ορισμένες από τις δηλώσεις που άκουσα δεν είναι μόνο ντροπιαστικέ, είναι και επικίνδυνες. Δυσχεραίνουν τα πράγματα αντί να οδηγήσουν σε μια κοινή προσπάθεια αντιμετώπιση των προκλήσεων. Σε ό,τι αφορά τα νούμερα που αναφέρονται, δεν μπορεί κανείς να ρίχνει στο ίδιο καλάθι διαφορετικά στατιστικά δεδομένα και να κάνει ένα συνονθήλευμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αλλά και αν ακόμα ήταν αλήθεια ότι ένας αριθμός εργαζόμενων θα εκτοπιστεί από άλλους που θα έλθουν, γιατί άραγε, τίθεται το ερώτημα, μήπως οι νέοι που θα έλθουν είναι καλύτεροι, καλύτερα εκπαιδευμένοι, έχουν καλύτερα προσόντα, τότε κάτι δεν πάει καλά με τα συστήματα εκπαίδευσή μας. Ή μήπω θα προτιμήσουν οι εργοδότες τους νέους διότι θα είναι διατεθειμένοι λόγω της κατάστασής τους να δεχθούν χαμηλότερα ημερομίσθια ή μισθου Τότε πάλι κάτι φταίει στο κοινωνικό μας σύστημα. Στην κοινωνική Ευρώπη, στη στρατηγική 2020. Εν προκειμένου, νομίζω ότι είναι εντελώς λάθος η συζήτηση εάν οδηγεί στον περιορισμό της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων, διότι αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο για τις αγορές εργασίας, αλλά διότι η πολιτική μας, με ομικρονιώτα δηλαδή, στις χώρες μέλη, δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έχουμε και μια αξιοπρόσεκτη εξέλιξη. Για τους δικούς μας απαιτούμε και τους λέμε ότι η ελεύθερη διακίνηση είναι κάτι το καταπληκτικό. Πολλοί νέοι θα έχουν καλύτερη μοίρα στην αγορά εργασία, εάν έχουν και εμπειρίε από την Ελλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή είμαστε υπέρ. Όταν όμω πρόκειται να έρθουν άλλοι στι δικέ μα χώρε. α, τότε όχι, να κλείσουμε τι πόρτε. Αυτά δεν γίνονται. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πραγματικά εδώ δεν έχουν καμία σχέση με την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, αλλά με το γεγονό περισσότερο ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε ξεκάθαρου κανόνε στην αγορά εργασία και να αντιμετωπίσουμε τη λεγόμενη μαύρη εργασία, να την εξαλείψουμε. Γι' αυτό το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να, να απευθύνω έκκληση να κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αφήσουν ελεύθερους τους εργαζόμενους. Τελευταίος είμαι εγώ προσωπικά. Πολύ σύντομα διότι οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες μίλησαν ξανά και ξανά. Ε, ας τα πούνε λιγάκι και οι Γερμανοί χριστιανοδημοκράτες. Όπως εγώ δηλαδή. Βέβαια όταν κανείς διευθύνει μια συζήτηση πρέπει να είναι αυτοσυγκρατημένος. Αλλά είναι σωστό. Δεν μπορούμε να εκτοπίζουμε μεν τους δε ή να θέτουμε μεν τους δε εκτός παιχνιδιού. Δεν είναι σωστό να γίνονται διακρίσεις. Όμως, εάν υπάρχουν κοινοί κανόνες και τηρούνται οι κοινοί κανόνες, 7 χρόνια μεταβατική περίοδος, ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής. Εγώ νομίζω ότι ήταν σωστή η εμπειρία αυτή. Πολλές από τις απειλές αυτές δεν υλοποιήθηκαν από τις απειλές που φοβόμασταν ότι θα υλοποιηθούν. Και αυτό είναι σημαντικό γεγονός. διαπιστώσαμε και το είπε ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι κανόνες που θεσπίστηκαν θα πρέπει να δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγκαιρα η αιτιολόγηση για ποιο λόγο γίνονται οι κανόνες αυτοί, για ποιο λόγο θεσπίζονται οι κανόνες και αυτοί και εφαρμόζονται. Και αυτά έγιναν βεβαίως σε σωστό χρονικό περιθώριο, δόθηκαν ενημερώσεις. Ορισμένες χώρες αποτελούν μαγνήτη για τους νέους εργαζόμενους. Αλλά ούτε εδώ υπάρχει καμιά εγγύηση ότι θα παραμείνει έτσι. Και εδώ μπορεί να προκληθούν πολλές αλλαγές. Και η ελκυστικότητα πολλών χωρών μελών μπορεί να μειωθεί. Για την ερώτηση κυρία Ζίπελ, ποιοι θα έλθουν. Ναι, πολλοί προσφέρονται να εργαστούν με τελείως άλλες συνθήκες. Και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση εκείνων οι οποίοι είναι βέβαια για μακρό χρόνο άνεργοι στις χώρες αυτές. Και αν το δει κανεί αυτό, ότι γίνεται η προσπάθεια τελικά να σπρώξουν το φτηνό εργαζόμενο κατά του ακριβού εργαζόμενου, τότε πρόκειται τελικά για μια κατάσταση ανασφάλειας. Εμείς όλοι είμαστε κατά της μαύρης εργασίας και βέβαια πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Ορισμένοι ζητούν κατώτατο μισθό. Εμείς λέμε στο δικό μου κόμμα να υπάρξει ένα κατώτατο όριο των μισθών που να θεσπιστεί και νομοθετικά. Λένε οι μεν που να το συμφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι, λέμε εμείς. Ανακλάδο, αναπεριφέρεια μπορεί να είναι διαφορετικό το όριο αυτό. Αυτό είναι ο ρόλο όμω των κοινωνικών εταίρων. Υπάρχουν βέβαια, όπω εξήγησα, κάποιε διαφοροποιήσει, κάποιε διακρίσει που έχουμε οι δύο πλευρέ, σοσιαλδημοκράτε και οι χριστιανοδημοκράτε. Όμω το βασικό στοιχείο είναι ότι δεν επιτρέπεται να γίνονται διακρίσει, δεν επιτρέπεται να γίνεται dumping, όπου τελικά να σπρώχνουμε του μεν, εργαζόμενου δηλαδή, κατά τον δε. Και ένα άλλο πράγμα θεωρώ σωστό δεν μπορούν να ερμηνεύονται τα γεγονότα ώστε να αποτελούν βάση για ιδεολογικούς αγώνες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Χρειαζόμαστε αγορές εργασίας που να λειτουργούν στη βάση εμπιστοσύνης. Ήδη στη δική μας Επιτροπή έχουμε πολλούς ε, θαυμάσιους συναδέλφους από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, των οποίων η συνεργασία είναι ανεκτήμητη και έχουμε νομίζω την σωστή βάση για να καταφέρουμε να αλλάξουν οι νοοτροπίες και στις χώρες μέλη. Εδώ λοιπόν τώρα εξαντλήθηκε ο κατάλογος ε, των εγγεγραμμένων αγορητών. Κύριε Μωράν, έχετε τώρα θαυμάσια ευκαιρία να μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας τέθηκαν, έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να καταλήψουν την αίθουσα αυτή εκανοποιημένη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα διάφορα σας σχόλια. Φυσικά θα τα αναφέρω και στον Επίτροπο Βάντορ. Πριν επανέλθω πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, ε, θα ήθελα απλά να αναφέρω ξανά ότι αυτά τα μεταβατικά μέτρα αποτελούν ουσιαστικά εξαίρεση για μια θεμελιώδη ελευθερία με χρονικό περιορισμό των 7 ετών που δεν μπορεί να παραταθεί Δηλαδή το αμετάκλητο τέλος αυτών των μεταβατικών μέτρων για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2013. Η πηγή αυτών των εξαιρέσεων ε, υπάρχει στην συνθήκη ένταξης, δηλαδή αυτή είναι η νομική βάση και εκεί έχουν προβλεφθεί οι τρεις φάσεις μαζί με το μηχανισμό ειδοποίησης για την είσοδο στην τρίτη φάση. Όσον αφορά το σχόλιο για την αξιολόγηση εκ μέρους μας ε, το τι συνέβη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άνοιξαν τις αγορές εργασίας τους στους Βουλγάρους και Ρουμάνους αυτή είναι μια αξιολόγηση που παρουσιάσαμε στην εκθέση του 2011 και σύμφωνοι με όσα είπα προηγουμένως ότι γενικώ ε, η οικονομική επιρροή ήταν θετική μετά από αυτό το άνοιγμα. Υπάρχουν κοινωνικές επιπτώσεις περιορισμένες κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τους ε, αμοιβέ και γενικώ ε, θετικές επιπτώσεις ε, για τη γενικότερη λειτουργία της αγοράς εργασίας για την κάλυψη των ενδεχομένων ελλείψεων εξειδίκευση. Τώρα, α περάσουμε στο πού βρισκόμαστε με τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο αυτή τη τρίτη φάση των μεταφατικών μέτρων. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας διαδικασίας ε, σε βάθος εξέτασης. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν ισχυρά επιχειρήματα τα οποία να συνοδεύουν τις ειδοποίησεις τους. Πρόκειται για μια περίπλοκη ανάλυση. Επειδή οι συνθήκες ένταξης αναφέρουν ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρήσουν μεταβεδικά μέτρα στην τελευταία φάση σε περίπτωση παρενόχλησης της αγοράς εργασίας τους ή κινδύνων παρενόχλησης της αγοράς εργασίας τους. Αυτές οι παρενοχλήσεις, αυτά τα προβλήματα δεν σχετίζονται απαραίτητα με την άφηξη των ε, Βουλγαρών και Ρουμάνων εργαζόμενων. Μπορεί να είναι γενικότερης φύσης ε, τα επιχειρήματα λοιπόν που προβάλλουν τα κράτη-μέλη. Είναι επιχειρήματα που μπορεί να αφορούν τη δική τους εκτίμηση της εξέλιξης της δικής τους οικονομικής εθνικής κατάστασης όσον αφορά την αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ειδοποίηση περιλαμβάνει ενημερωτικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση της αγοράς εργασίας σε εθνικό επίπεδο και που σχετίζονται επίσης με τις ε, ίδιες οικονομικές προοπτικές του κάθε κράτους που πραγματοποιεί την ειδοποίηση. Ειδικότερα οι προβλέψεις ανάπτυξης, ε, οι προβλέψεις απασχόλησης, ε, ενδεχομένως επιδίνωσης ή όχι της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία δεν είναι τα ίδια προφανώς για κάθε κρατός που βασίζονται σε κάποιο βαθμό σε εκτιμήσεις διότι υπάρχουν φυσικά βασίζονται σε αναλύσεις οι οποίες θεμελιώνονται σε, βασίζονται σε κάποιες οικονομικές υποθέσεις αυτό που έκανε η Κομισιόν καλώντας μια σειρά κρατών μελών ε, να ε, συμπληρώσουν με κάποιες πληροφορίες τις εξηγήσει τους ήταν το να βεβαιωθεί, προσπαθούσε δηλαδή η Κομισιόν να βεβαιωθεί ότι η ανάλυση που γίνεται όσον αφορά την κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις προοπτικές εξέλιξεις των αγορών εργασίας βασίζεται όντως σε αντικειμενικά επιχειρήματα, σε σαφείς αριθμούς και σε υποθέσεις με τις οποίες μπορούμε να συμφωνήσουμε, δηλαδή να οδηγήσουμε τα κράτη-μέλη σε μια ε, ικανή, σωστή αιτιολόγηση, αξιολόγηση της αγοράς εργασίας τους εν των κινδύνων παρενόχλησης ε, της αγοράς εργασίας, ε, κινδύνων γενικής φύσης. Το σκεπτικό επίσης είναι να διατηρηθεί αυτός ο άλγος με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ενδιάμεση αξιολόγηση για την επαναξιολόγηση αυτών των συνθήκων, οι οποίες μπορεί να εξελίσσονται μέσα στα ε, χρόνια, ειδικότερα εντός του 2013. Και έτσι τα κρατημέλη να χρειαστεί να επανεξετάσουν τις θέσεις τους όσον αφορά εξελίξεις ενδεχόμενες στις αγορές εργασίας. Αυτή είναι η ουσία των ανταλλαγών που έλαβαν χώρα και αυτή είναι η ουσία των αναλύσεων της Κομισιόν, του, ε, του, του τρόπου με τον οποίο η Κομισιόν αναλύει αυτές τις πληροφορίες που τις παρέχουν τα κρατη Δηλαδή η Κομισιόν προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι διάφορες υποθέσεις ε, για την αγορά εργασία στα διάφορα κράτη-μέλη ε, είναι πράγματι ε, σωστές και εύλογες και αντιστοιχούν και στις δικές μας υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, για να δώσω τις απαραίτητες απαντήσεις, εδώ μιλάμε για μια παρακολούθηση η οποία θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι ενδεχόμενε αλλαγέ κατάσταση τη αγορά εργασία στα κράτη που έχουν διατηρήσει του περιορισμού θα μπορέσουν να ε, ενσωματηθούν και να αποτελέσουν το αντικείμενο εξέταση ε, μαζί με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μωράν και για το μήνυμά σας ότι θα γίνει μια ενδιάμεση επανεξέταση. Μίλης μόνο ότι έχουμε και άμεση μετάδοση των ε, συνεδριάσεων μας σε αντίθεση με άλλα κοινοβούλια. Είναι σημαντικό λοιπόν το μήνυμα που περνά και από το διαδίκτυο καθώς συνεδριάζουμε και ενδιαφερόμενοι μπορούν να μας παρακολουθούν. Μπορώ, νομίζω ότι είναι θετικό το μήνυμα αυτό, έστω και αν υπάρχουν εδώ δυσκολίες. Το 19 τώρα, ο ρόλος της εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Η ε, κυρία Χιουσμένοβα από τη Βουλγαρία θα μπορέσει να λάβει το λόγο για να εξηγήσει την γνωμοδότησή της. Ελπίζω πολύ η γνωμοδότηση αυτή να βρει απήχηση στην Περιφερειακή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη, ώστε και οι σκιώδεις ε, εισηγητές ε, να μπορέσουν να τοποθετηθούν. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Είναι πολύ κατάλληλη στιγμή που έτυχε να παρουσιάζουμε αυτή την ε, έκθεση γιατί συμπίπτει και με την πρόταση για την πολιτική συνοχή για την περίοδο 2014-2020. Προσπαθούμε στην ε, γνωμοδότηση αυτή να παρουσιάσουμε τις βασικές εξελίξεις στον τομέα τη εδαφική ε, ανάπτυξη και στον τομέα τη ε, κοινωνική συνοχή. και με ποιον κατάλληλο μηχανισμό μπορούμε να βελτιώσουμε την καλύτερη ανάπτυξη των υπηρεσιών, την καλύτερη εκπαίδευση, υγεία και τη μείωση τη φτώχεια που είναι από του βασικού στόχου της στρατηγικής 2020. Σε αυτό το πλαίσιο, να πω ότι η δαφική προσέγγιση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που προβλέπει το Ταμείο είναι κάτι πολύ σημαντικό για να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό όμως θα γίνει αν υπάρχει το κατάλληλο δυναμικό στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι όταν μιλώ για δυναμικό δεν αναφέρω μόνο στο διοικητικό δυναμικό, αλλά και στο δυναμικό των κοινωνικών εταίρων που θα πρέπει να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των πολιτικών. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε τα προαπαιτούμενα, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε πρακτικά την εδαφική προσέγγιση και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης και να προχωρήσουμε περαιτέρω στον τομέα της ε, συνοχής επίσης να πω ότι έχουν δρομολογηθεί σχετικές συμφωνίες ε, εταιρικής σχέσης για, την, ε, τα υπηρεσιακά προγράμματα και εν προκειμένου είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί φωνή όλων των ενδιαφερομένων μερών για να υπάρχει συμπερίληψη όλων των τοπικών φορέων και να μπορέσει να οικοδομηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Τα υπηρεσιακά προγράμματα θα πρέπει να βασίζονται στην εις ανάλυση του δυναμικού που υπάρχει για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και οι ολοκληρωμένες στρατηγικές θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά στις γεωγραφικές περιφέρειες, ιδίω περιφέρειες εκείνες που αντιμετωπίζουν περισσότερο το πρόβλημα της ανεργίας. Έπειτα υπάρχουν ομάδες στόχοι που έχουν επηρεαστεί χειρότερα από το πρόβλημα της εκδικής μεταχείρισης και της έλλειψης ενσωμάτωσης. Εκεί λοιπόν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο συνεχίζουμε να είμαστε μάρτυρες ε, τεράστιων ανισοτήτων στον κοινωνικό τομέα και και μιλάμε για ανισότητε, όχι μεταξύ περιφερειών μόνο, αλλά και μέσα στις ίδιες περιφέρειες. Γι' αυτό θα πρέπει να καταρτιστούν προγράμματα που να μπορούν να ανταποκριθούν στι περιφερειακέ και υποπεριφερειακέ ανάγκε. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να συνεχίζει να υποστηρίζει την ανάπτυξη τοπικών προσεγγίσεων για την απασχόληση και την κοινωνική ε, συμμετοχή. Στην γνωμοδότησή μου δεν κατάφερα να συμπεριλάβω και τις υποπεριφερειακές ε, στρατηγικές που μπορούν να ενθαρρύνουν ε, την κινητικότητα των νέων, τα δημοκρατικά στοιχεία κτλ. Όμως θα κάνω μια σχετική πρόταση ε, με τη μορφή τροπολογιών για αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω σε μια συζήτηση για τις δικές σας προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ιουσμένοβα. Φρεντερίκ Ντάρνταν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε η συγκήτρια, η γνωμοδότηση αυτή, συμφωνώ και εγώ, είναι επίκαιρη και συμπληρώνει τις συζητήσεις μας για τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία και τους κανονισμούς και την διάρκειά τους και την θέση τους μέσα στα δημοσιονομικά και βεβαίως μέσα στο πλαίσιο του ε, πρόσεχους δημοσιονομικού πολιτούς ε, προγράμματος. Είναι σαφές ότι ο ρόλος της ε, εδαφικής ανάπτυξης είναι κέριος. Και η ορατότητα των προγραμμάτων στο τοπικό επίπεδο είναι σημαντική και οι τοπικές αρχές πρέπει να παίζουν ένα ρόλο σε συνεργασία με τους διαφόρους φορείς της πολιτικής συνοχής. Πριν όμως εκφράσω άποψη για το σχέδιο ε, γνωμοδοτήσεως, θα ήθελα να τονίσω πρώτα ότι είναι απαραίτητο να οριστεί η έννοια, διότι μιλούμε για δαφική ανάπτυξη και υποθέτω ότι μέσα στην έκθεση, στην γνωμοδότηση δηλαδή, τη συναδέλφου μας θα περιληφθεί και ένας ορισμός και στον ορισμό αυτό θα μπει και αυτό το κοινωνικό στοιχείο της ε, εδαφικής ανάπτυξης. Τώρα, το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που μας έχει υποβληθεί επαναλαμβάνει ορισμένα θετικά ε, πράγματα και αποτελεί μια καλή βάση για περαιτέρω εργασία, ιδίως για το θεμελιώδη χαρακτήρα της εδαφικής ανάπτυξης μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Άλλο στοιχείο που είναι η αναγκαιότητα να προσαρμόζονται τα προγράμματα στις περιφερειακές και τοπικές συνθήκες με λήψη υπόψη της αρχής της επικουρικότητας. Και εδώ θα ήθελα να ακούσω από την εισηγήτρια ορισμένα πιο συγκεκριμένα για την παράγραφο 3 που αναφέρεται στο θέμα αυτό. Επίσης, οι τεχνικές πτυχές των συμβάσεων μεταξύ ευρωπαϊκών οργάνων και τοπικών φορέων και ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα μέρη που ενδιαφέρονται για την εκτέλεση των συμβάσεων. Είναι λοιπόν ορισμένα σημαντικά πράγματα τα οποία περιλαμβάνει η έκθεση γνωμοδοτήσεως και που ανταποκρίνονται στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και εμείς. Θα μου επιτρέψει η συγγήτρια να ε, υποβάλω ορισμένε τροπολογίες και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία για παράδειγμα την ανάγκη να ρηχθεί φως στο ρόλο των τοπικών αρχών για την πλοπή στρατηγικής 2020, για τη μείωση της φτώχειας, κάτι το οποίο αναφέρθηκε και στην έκθεση για την πλατφόρμα για την ε, καταπολέμηση της φτώχειας. Σε ό,τι αφορά τα ενδιαφερόμενα, τους ενδιαφερόμενους φορείς πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιοι είναι και πώς θα συμμετάσχουν, κυρίως οι κοινωνικοί εταίροι. Επίσης η Κομισιόν έχει κάνει πρόσφατα ορισμένες ανακοινώσεις σχετικά με την εφαρμογή του Κοινωνικού Ταμείου για την καταπολέμηση της ε, φτώχειας, της ανεργίας των νέων, αλλά βέβαια οι δράσεις αυτές παραμένουν ασαφείς καμιά φορά και θα έπρεπε ίσως να τονιστεί η ανάγκη να διευκρινιστούν, να γίνουν πιο ξεκάθαρες. Και τέλος στο επίπεδο της αναθεωρήσεως, στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής δηλαδή, είναι σημαντικό νομίζω να επεκταθεί η πολιτική αυτή στο σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας. Είναι και, ε, ε, υπάρχει και ο προβληματισμός των ενδιάμεσων περιφερειών και όπως ε, φάνηκε στην έκθεση ΠΠΕΡ και είναι σημαντικό να περιληφθεί το στοιχείο αυτό και σε τούτην εδώ τη γνωμοδότηση ώστε να είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να καλυφθεί όλη η Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Αυτά λοιπόν είναι κάποια πρώτα στοιχεία που ε, θέλω να συμβάλλω στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ Φρεντερίκ. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Συγήτρια, λοιπόν, αν θέλετε να απαντήσετε στα σχόλια του κυρίου Ντάρντεν. Merci euh, pour le commentaire du collègue. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο του συναδέλφου. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα γαλλικά. Φυσικά το σχέδιο που παρουσίασα δεν είναι το τελικό. Γι' αυτό το λόγο τα όποια σχόλια, προτάσεις, ιδέες ε, των συναδέλφων μου που είναι σκιώδεις εισηγητές ε, θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμα για μένα θα με βοηθήσουν να, να δώσω μια οριστική μορφή στο κείμενο, να είναι πιο ισορροπημένο και πιο ολοκληρωμένο. Φυσικά θα μπορούσα να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, των συναδέλφων ενδεχομένως στο τέλος όταν το κείμενο θα είναι έτοιμο. Αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι για να έχουμε μια πιο αποτελεσματική πολιτική ε, συνοχής θα χρειαστεί να βελτιώσουμε τις ικανότητες όλων των εταίρων. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τελικά ένα πιο ολοκληρωμένο κείμενο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσει όλων των εταίρων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι 3η Μαΐου, 3η Πέμπτου, στις 12 το μεσημέρι. Θα σας κακοσυνηθήσουμε βεβαίως, διότι θα αλλάξουμε πάλι τώρα πρόεδρο και θα ακολουθήσει ο κ. Φιλίπ Μπουλάν ως ομιλητής. Καλησπέρα σε όλου. Είναι η πρώτη φορά που προείσταμε μία συνεδρία σε επιτροπής μας. Ελπίζω να μην κάνω κάποιο λάθος. Αν όμω το κάνω, σας ε, παρακαλώ τουλάχιστον να έχω την κατανόησή σας. Ας περάσουμε στο σημείο 20 τη διάταξης για τον προπολογισμό του 2013, εντολή για τον ε, τριμερή διάλογο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φιλίπ Πουλά, ο οποίος είναι συντάκτης της γνωμοδότησης που είναι υποσύζητηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συναδέλφοι, θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση του τι προτείνουμε για τον προπολογισμό του 2013. Κατά την άποψή μου η Ευρώπη καταφέρει να αφιερώσει όλες τις δυνάμεις για να προωθήσει μια οικονομική διακυβέρνηση και πρέπει να δώσει τις ίδιες διανάμεις για μια κοινωνική διακυβέρνηση. Αυτό θα βασιστεί σε ενέργειες που ευνοούν την, συνοχή και την κοινωνική συνοχή. Τα κονδύλια που χρησιμοποιεί η Κομισιόν είναι αφιερωμένα στην δίωξη αυτών των στόχων. Ο προπολογισμό του 2013 θα πρέπει να υποστηρίξει τι εμβληματικέ πρωτοβουλίε όπω την κοινοτομία. Ωστόσο, ο προπολογισμό του 2013, παρότι είναι ο τελευταίο για το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν πρέπει να περιοριστεί στη ε, κονδυλία για τα προγράμματα που, των οποίων η εκτέλεση ολοκληρώνεται πρέπει να προωθήσει μια δυναμική για να βοηθήσει όσου νέους αναζητούν εργασία και για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να επαναξιολογηθεί και να αναδρομολογηθεί για το 2014-2020 όπως παρουσιάστηκαν οι προοπτικές από την Κομισιόν ε, πέρυσι πρέπει να έχει ένα πιο ευρύ πεδίο διότι οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο θα είναι επιλέξιμες πλέον για υποστήριξη του κοινωνικού ταμείου και μεγαλύτερη σημασία θα δοθεί στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων πρότασή μου είναι να μην περιμένουμε το 2014 για να καταπολεμήσουμε την ενέργεια των νέων. Είναι αρκετά κρίσιμη η τρέχουσα κατάσταση ώστε από τώρα να εφαρμοσουμε όλα τα μέτρα που θα επιτρέψουν τη μείωση της ενεργείας και ειδικότερα των νέων. Ξέρω ότι έχουμε περιορισμούς δημοσιονομικούς, ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν μπορούν να είναι απεριόριστες, αλλά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για τον προπολογισμό του 2013 για να περάσουμε ένα σημαντικό μήνυμα ώστε να βοηθήσουμε όσο αναζητούν εργασία. Αυτό πρέπει να το κάνει η δική μας Επιτροπή. Επίσης πρέπει να υποστηρίξουμε την προσαρμογή ε, των ικανοτήτων στους τομείς που, όπου υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, να βοηθήσουμε τη μικροχρηματοδότηση χωρίς να ξεχνάμε το ΙΡΕΣ, το οποίο βοηθά και ενθαρρύνει όλες τις ε, πρωτοβουλίες που βοηθούν τις προσλήψεις σε τοπικό επίπεδο και στα σημεία που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Επίσης, οι δράσεις για την καινοτομία και για κοινωνική πρόοδο που αναλαμβάνουν οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να χαίρουν μια ε, οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ είναι οι προτεραιότητε που θα ήθελα να αναπτύξουμε στο ψήφισμα που σα προτείνω. Φυσικά παραμένω στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε προτάσεις και από εσάς και από τους συναδέλφου σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε εισηγητή. Έχουμε έναν συνάδελφο που έχει εγγραφεί. Μπορείτε να ζητήσετε λοιπόν το λόγο κατά την ομιλία του. Δίνω το λόγο στον κύριο Νταρντέν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα λόγια σε σχέση με αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης Απλά για να πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνώ με το σχέδιο γνωμοδότησης που υποβάλλει ο συναδελφός Φιλιμπουλό. μια καλή αφετηρία για συζητήσεις. Θα αναφέρω κάποια σημεία που μου φαίνονται ενδιαφέροντα στο σχέδιό του, ειδικότερα την ανάγκη κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 2020. Πιστεύω ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να υπενθυμίζουμε, ειδικότερα όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας και της ανεργίας των νέων ε, το γεγονός ότι επισημαίνουμε το ρόλο των ε, κοινωνικών εταίρων, τη χρήση του Ταμείου ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ειδικότερα για τον επαναπροσανατολισμό στους τομείς του μέλλοντος, την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικά θέματα, την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και την εφαρμογή ε, συνθήκων κατάλληλων εργασίας ε, για ε, κατάλληλων για τους πολίτες μας αναφέρεται και εδώ στην Επιτροπή μας και στο πλαίσιο των εργασιών μας και των τροπολογιών που θα υποβάλουμε θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε κάποια θέματα όπως πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βρούμε καλύτερη χρηματοδότηση, επαρκή χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες, ε, τις εμβληματικές πρωτοβουλίες, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο όσον αφορά τον ορισμό του της επαρκούς χρηματοδότησης. Επίσης όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέσα που αφιερώνονται στις πρωτοβουλίε τη Κομισιόν για την απασχόληση των νέων θα πρέπει να αναφέρεται καθαρά είναι σημαντικό να ζητήσουμε τι σχετικέ πληροφορίε από την Κομισιόν ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε τη σπουδαιότητα αυτή τη ε, πρωτοβουλία. Όσον αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε κάπως να συμπληρώσουμε, να ενισχύσουμε τη θεματολογία, ώστε να υποστηρίξουμε αυτό το εργαλείο που μου φαίνεται σημαντικό. Μερικές φορές επιμένουμε, ειδικότερα στο Συμβούλιο, στο γεγονός ότι ότι δεν ε, δαπανώνται επαρκώς ε, τα κονδύλια Ωστόσο βλέπουμε ότι δεν έχουμε αρκετές ε, χρηματοδοτικές πιστώσεις και χρειάζεται να κάνουμε μεταφορές. Είναι πως μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό στον προπολογισμό να έχουμε επαρκείς πιστώσεις ε, όσον αφορά τα εμβληματικά προγράμματα και θα μπορούσαμε να κάνουμε και προτάσεις για προσθήκη εμβληματικών προγραμμάτων που εγώ θεωρώ σημαντικά. Πιστεύω επίσης ότι η χρηματοδότηση για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων θα μπορεί να συσχετιστεί και με τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. Επίσης, όταν επιμένουμε στη σπουδαιότητα των πιστώσεων πληρωμής στο πλαίσιο του προπολογισμού του 2013, γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν προσέχουν ειδικότερα για αυτό το θέμα και ειδικότερα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις του προπολογισμού 2012 είχαμε ανεπαρκή επίπεδα πιστώσεων για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτές τις πολιτικές συνεπώς θα πρέπει να επιμείνουμε λίγο παραπάνω σε αυτό το σημείο αυτά είναι μερικές δικές μου προτάσεις και εκτιμήσεις ευχαριστώ ε, Ευχαριστούμε πολύ λέει η Προεδρεύουσα Άλλος κανείς δεν μου έχει ζητήσει το λόγο. Επιθυμεί κάποιος να παρέμβει για το θέμα αυτό. Πριν δώσω το λόγο πάλι στον εισηγητή. Η Κομισιόν. Από ό,τι φαίνεται δεν επιθυμεί. Άλλες παραμβάσεις δεν διαγράφονται στον ορίζοντα. Ο κύριος Μπουλάου. Ευχαριστώ τον κύριο Νταρντέν για τις προτάσεις του, άλλωστε με βρίσκουν σύμφωνο. Προφανώς η σταδιακή 2020 πρέπει να αποτελέσει το στόχο μας. Οι προτάσει που κάνω είναι περισσότερο γενικέ, είναι περισσότερο κατευθύνσεις. Ο κύριος Νταρντέν νομίζω θα χαρεί να δει ότι συμφωνούμε στα περισσότερα από τα όσα τόνισε και σε μια άλλη έκθεση της κυρία Στάινμπρικ όπου είμαι εισηγητής από την πλευρά του Λαϊκού Κόμματος όπου τίθεται όλα αυτά τα θέματα για παράδειγμα τα πιλωτικά προγράμματα και οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις που πρέπει εκεί να προωθηθούν ως ιδέες και για το ΦΕΜ δηλαδή εννοώ το Ταμείο προσαρμογή στην κοσμιοποίηση καθώς και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Υπάρχει μια σύγκληση μέσα στις εκθέσεις αυτές και στην εργασία μας. Δεν υπάρχουν νομίζω μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις προσεγγίσεις μας, τουλάχιστον σήμερα. Σημείωσα τις σκέψεις που εξέφρασε και επαναλαμβάνω την διαθεσιμότητά μου και προς τις άλλες και άλλους ευρωβουλευτές για το θέμα του προϋπολογισμού για την εργασία που θα επανέλθουμε όταν θα μας υποβάλει πρόταση η Επιτροπή Προϋπολογισμών πιο συγκεκριμένη. Σε μια προσπάθεια να οργανωθούμε θέμα όπως τα εξηγήσατε και εσείς κύριε Νταρδέν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουλάν. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 27η Απριλίου. Την Παρασκευή δηλαδή έως τις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο είναι η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας. Όμως η γήτρια δεν είναι παρούσα, οπότε προτείνω να πάμε στο σημείο 22 και μετά θα επιστρέψουμε στο σημείο 21. Το σημείο 22 είναι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013-2017 που εισηγητής είναι ο κύριος Άνταμ Κόσα, στον οποίο δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου η χαρά με την οποία θα συνοψίσω ε, τις τροπολογίες. Δεν ήμουνα έτοιμος να πω την αλήθεια, ε, γιατί περιμένω ακόμη αυτό που υπέβαλαν τροπολογίε για να κάνουμε τη συζήτηση. Δεν ξέρω πώ να κάνουμε τη συζήτηση. Βλέπω έναν από του σκιώδει εισηγητέ να είναι εδώ παρόν, αλλά θα ήθελα όλου να είναι παρόντε στη συζήτηση. Σε μια χρονική στιγμή προσπαθούμε να θεσπίσουμε προτεραιότητε για το στατιστικό πρόγραμμα, είναι καλό να κάνουμε μια στις επί της ουσίας. Πρόεδρε, τι λέτε, μήπως να κάνουμε μια παύση αυτή τη στιγμή, να συνεχίσουμε αργότερα. The problem is Επιλύθηκε το πρόβλημα, λέει η Πρόεδρος. Μια στιγμή, κυρία Ράπτη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ε, μπήκατε στην αίθουσα. Η συγγήτρια του σημείου 21, θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας. Παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Αν είναι έτοιμη η συγγήτρια, παρακαλώ να σας δώσω αμέσως το λόγο. Κυρία Σιλβάνα Ράπτη έχει το λόγο. Ε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη καταρχήν και από εσά και από όλους τους παρευρισκόμενους αλλά είχα προγραμματίσει διαφορετικά με βάση την ημερήσια διάταξη α, της α, δουλειές μου. Συγγνώμη και πάλι και προχωρώ. Λοιπόν, ε, μιλάμε για μία γνωμοδότηση που έχει να κάνει με την αναθεώρηση του κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας. Ε, με λίγα λόγια, τι είναι αυτό το θέμα. Το 2004 γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και ένας μηχανισμός για να στηρίξει αυτή την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Πολύ σοφά σκεπτόμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει και ξέρουμε όλοι μας ότι για να είμαστε καλά στο σπίτι μας πρέπει να είναι καλά και όλη η γειτονιά μας. Άρα για να μπορεί να είναι σε ειρηνικό, δημοκρατικό και περιβάλλον με ευημερία η Ευρώπη, έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε δημοκρατικούς θεσμούς, ειρήνη και ευημερία και στις χώρες τις γειτονικές. Οι χώρες αυτές οι γειτονικές είναι 16. Και βέβαια πρέπει να σημειώσω ότι το 2004 όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και ο μηχανισμός της ε, δεν είχαν συμβεί όσα έχουν συμβεί στο μεταξύ στο τόξο αυτό που λέμε της Αραβικής Άνοιξης. Καθώς ο μηχανισμός αυτός μπήκε σε λειτουργία, όπως συμβαίνει με όλους τους μηχανισμούς, διαπιστώθηκαν ε, κάποια προβλήματα. Ε, ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε, να γνωμοδοτήσουμε σε σχέση με αυτό το μηχανισμό έχοντας στο μυαλό μας, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, δύο πράγματα. Πρώτον, ο μηχανισμός αυτός να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός και δεύτερον, να μπορούμε η βοήθεια την οποία προσφέρουμε να είναι περισσότερο συγκεκριμένα στόχευμένη και το κυριότερο να φτάνει έγκαιρα στους γειτονές μας εκεί που πρέπει. Α, στο ρυθμό. Μιλάω πολύ γρήγορα μου λένε. Οκ. Πηγαίνω πιο σιγά. Λοιπόν, η σημερινή γνωμοδότηση είναι στην ουσία συνέχεια μιας γνωμοδότησης που είχαμε κάνει σε αυτήν εδώ την Επιτροπή πριν από μερικούς μήνες. Ήταν μια γνωμοδότηση, παύλα, γνωμοδότηση πρωτοβουλίας που ερχόταν να κουμπώσει, να ταιριάξει με την έκθεση που γίνεται από την ΑΦΕΤ. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα στην νομοθετική γνωμοδότηση και πρέπει να δούμε μερικά πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Η δική μου προσέγγιση έχει να κάνει κυρίως με τα κοινωνικά θέματα με τα κριτήρια σε σχέση με τα κοινωνικά θέματα στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας που αισθάνομαι ότι δεν θίγονται τόσο όσο θα έπρεπε. Ε, μέσα στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας είναι οι παρατηρήσεις και οι τροποποιήσεις που προτείνω. Ανάμεσα σε αυτά σημειώνω και την φιλοσοφία του νέου κανονισμού, μια φιλοσοφία που λέει ότι να δίνουμε περισσότερη χρηματοδότηση σε όσους επιδεικνύουν καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. More for more. Ε, θεωρώ πως πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, αλλά ε, θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους, υπογραμμίζω, ως προϋποθέσεις για την οικονομική ενίσχυση. Ε, σας λέω πολύ σύντομα ε, τις τρεις ε, έτσι, ε, πώς να το πω, τις τρεις βασικές αρχές που έχω στο μυαλό μου όταν προτείνω τις τροπολογίες. Η πρώτη αρχή είναι τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Η δεύτερη είναι η κοινωνική προστασία και κοινωνική δικαιοσύνη και η τρίτη είναι βέβαια η απασχόληση. Ε, πιο συγκεκριμένα ζητώ και προτείνω και ασφαλώς θέλω τη γνώμη όλων σας ε, και των ε, σκιωδών και όλων των συναδέλφων ένα κανονιστικό πλαίσιο για θέματα κοινωνικής προστασίας. Ζητώ επίσης να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, να βελτιωθούν οι πολιτικές απασχόλησης και μέσα σε αυτές να συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα εκπαίδευσης και τα προγράμματα κατάρτισης Ζητώ να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και βέβαια να αντιμετωπίζονται οι καταχρήσεις στην αγορά εργασίας. Θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να εφαρμόζονται τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Δίνω ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο της λεγόμενης κυκλικής κινητικότητας που ξέρουμε όλοι ότι επιτρέπει να αποκτώνται γνώσεις, να αποκτάτε τεχνογνωσία, αλλά παράλληλα η γνώση αυτή πρέπει να επιστρέφει στον τόπο που έχει ανάγκη. Επίσης, θέλουμε καλύτερη αντιστήχηση των δεξιοτήτων με τη ζήτηση εργασίας. Και τέλος, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα, πρέπει να είναι υποχρεωτική, έτσι το θεωρώ εγώ, η δυνατότητα να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών στον κοινωνικό διάλογο και στη διαβούλευση προκειμένου να θεσπίζεται νομοθεσία. Εδώ βάζω μία τελεία. Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας και περιμένω πραγματικά με ανυπομονησία, επιτρέψτε μου την έκφραση, ε, τις παρατηρήσεις σας, τις υποδείξεις σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά γίνεται για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χολοκόφσκι έχει ζητήσει το λόγο μόνο έως τώρα. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλος αγορτής. Παρακαλώ, αν επιθυμείτε να πάρετε το λόγο, να μου κάνετε ένα σήμα. Ο κύριος Χολοκόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Θέλω να ευχαριστήσω την αγαπητή συνάδελφο Σιλβάνα Ράπτη για αυτή τη γνωμοδότηση Είμαι μονίμος συγητή στην Επιτροπή Προπολογισμών για αυτό το μέσο και θα ήθελα να μοιραστώ κάποιε παρατηρήσει ε, που παρουσίασα και στη δική μου έκθεση. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι η πρόταση της Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Μεσογειτονίας ε, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δημιουργούνται προϋποθέσεις για πιο αποτελεσματική υποστήριξη και πιο ταχεία. Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν θα είναι πιο απλός και πιο εύχριστος. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Δεύτερον, υποστηρίζω την αρχή για την οποία μιλήσε η αξιότιμη κυρία Ράπτη, το είναι αρχή more for more. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να καθορίσουμε σαφή διαφανή κριτήρια και αντικειμενικά κριτήρια για την εφαρμογή αυτού του κριτηρίου. Τέλο, πιστεύω ότι οι γειτονικέ χώρε θα πρέπει να υποστηριχθούν ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν του θεσμού του ώστε να μπορέσουν να εγγυηθούν την κατάλληλη αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων, ώστε να βελτιωθεί επίσης η προστιθέμενη αξία. Πρέπει να συνδεθεί αυτό ο μηχανισμός με τα άλλα, ε, με τους άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Σκέφτομαι την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την ΠΕΡΣ. Σκέφτομαι για τα εναλλακτικά ταμεία για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ αυτού του μηχανισμού και των υπολείπων ταμείων. Θα πρέπει ωστόσο να αποφύγουμε την επικάλυψη μεταξύ αυτών των ταμείων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια συνεργασία μεταξύ αυτών των ταμείων. Επίσης είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική στην οποία θα συμμετέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεδομένου ότι προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας και είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη, για την οικονομική ανάπτυξη μάλιστα. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη αυτών των ε, επιχειρήσεων στις ε, γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για μεγαλύτερη οικονομική εφορία. Υπογραμμίζω επίσης το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχεδιασμό των χρηματοδοτήσεων για τα εθνικά προγράμματα και για τα διεθνή προγράμματα. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα αναστολής αυτών των χρηματοδοτήσεων εφόσον καταστεί απαραίτητο. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω αν θέλει κανείς άλλος ε, το λόγο, παρακαλώ. Κασίν. Ο κύριος Κασίν. Dear Chair, dear... Κυρία Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Συγήτρια, κύριε Ράπτη, κύριε συνάδελφοι, πριν από κάποιο διάστημα είχαμε συζητήσει και πάλι την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία πάλι με την ίδια συγγετρία. Και θεωρώ ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι μια λογική συνέπεια των συμπερασμάτων στα οποία είχαμε καταλήξει τότε. Το ίδιο πολιτικό μήνυμα θα ήθελα να περάσω. Η ευρωπαϊκή απασχόληση, και κοινωνικά πρότυπα, η απασχόληση, η ισότητα και η κινητικότητα είναι οι λέξεις κλειδιά. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το εργαλείο μπορεί να ανταποκριθεί ισότιμα στις διάφορες δημογραφικές τάσεις και στις διάφορες ανάγκες των δύο διαστάσεων της πολιτικής γειτονίας, την Ανατολική και την Μεσογειακή. Επίσης θα πρέπει να εμείνουμε στο εξή ότι αυτό είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Γι' αυτό να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το σχέδιο γνωμοδότησή σας και την κατεύθυνση προς την οποία κινείστε λίγες ε, ουσιαστικές αλλαγές, ε, διαφορές υπάρχουν μεταξύ μας. Όμως ε, έως την Πέμπτη το μεσημέρι θα λάβετε και τη δική μας γραπτή συμβολή εν προκειμένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρωτώ και πάλι αν θα ήθελε κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Ναι, ναι, θα σας δώσω αμέσως, κυρία Συγγήτρια, το λόγο να κάνετε τις τελευταίες παρατηρήσεις. Η Συγγήτρια. Κυρία Πρόεδρε, όλο μου δίνετε το λόγο και όλο εγώ ή δεν είμαι εδώ ή άλλα σκέφτομαι. Ε, λοιπόν, ε, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους για τις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις που έκαναν. Ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και το θέμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία και έχετε απόλυτο δίκιο στο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως επίσης και στο τρίτο σημείο που θίξατε, να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη. Ε, τώρα, στα άλλα ζητήματα που έβαλε, ο κύριος Κασίν είναι το, το θέμα της ανατολικής γειτονίας, να το πω έτσι, και το θέμα της μεσογειακής γειτονίας. Ε, υπάρχουν λεπτά λεπτές, να το πω έτσι, λεπτές αποχρώσεις. Δηλαδή, στη Μεσόγειο, το είπα και στην αρχή, δεν υπήρχε τίποτα από αυτήν την κατάσταση που υπάρχει σήμερα που ξανασυζητάμε την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Δεν υπήρχε τίποτα από αυτό το 2004 όταν γεννήθηκε αυτή η πολιτική. Άρα θα πρέπει να, να, να ζυγίσουμε κατά κάποιο τρόπο ε, το πώς θα μοιράσουμε την βοήθειά μας προς Ανατολάς και στη λεκάνη της Μεσογείου. Ε, είναι λέξη κλειδί το θέμα της ισοτιμίας. Αλλά η ισοτιμία μπορεί να έχει ε, διαφορετικές διαστάσεις. Παράδειγμα, ισοτιμία δεν είναι κατά τη δική μου γνώμη να δώσω 100 σε όλους. Θα πρέπει το ποσό που θα δώσω να μπαίνει σε μία κριτική εξέταση ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε γειτονική χώρα, ένα, και δεύτερον, ανάλογα στο τι προσδοκά η Ευρωπαϊκή Ένωση από την καλή γειτονία να το πω έτσι, με την χώρα αυτή ή με τις χώρες αυτές. Προς Θεού δεν θέλω να παρεξηγηθώ, θέλω ε, να, να γίνει σαφής η διάθεσή μου και πρόθεσή μου να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα κριτήρια, όλες τις παραμέτρους και να είμαστε πραγματικά δίκαιοι, έχοντας στο μυαλό μας ότι για μας παίζει τεράστιο ρόλο το να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, να προστατεύονται τα κοινωνικά δικαιώματα και η δημοκρατία με όλη τη σημασία της λέξης. Οι παρατηρήσεις που έκαναν οι συνάδελφοί μου ε, αισθάνομαι ότι με βοηθούν πάρα πολύ στην δουλειά αυτή που έχουμε να κάνουμε όλοι μαζί. Και βέβαια, ως την Πέμπτη που λύγει η προθεσμία για τις τροπολογίες, ε, περιμένω να δω τις τροπολογίες σας και εάν μπορέσουμε να συνυπογράψουμε και μαζί κάποιες από αυτές ή ενδεχομένως και όλες. Ε, ευχαριστώ και πάλι. Καλώς σας ευχαριστώ και εγώ. Όπως είπε και η διασηγήτρια, θα το επαναλάβω και εγώ, να μην το ξεχάσουμε, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών για αυτή τη γνωμοδότηση είναι 26 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Μεθαύριο λοιπόν, τώρα θα δώσω τη σκητάλη στην κυρία Σρότερ να ε, προεδρεύσει. Η κυρία Σουρέτερ, ευχαριστώ πολύ. Μα μένει ένα τελευταίο θέμα τη ημερησία διατάξεω, που είναι το υπαριθμόν 22, με θέμα Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013 έως 2017. Και η συγητής είναι ο κύριο Άνταμ Κόσα. Άνταμ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μία σύνοψη και να ζητήσω συγγνώμη γιατί ήμουν απόν στην τελευταία συνεδρίαση όταν συζητήθηκε η γνωμοδότηση. Ο συνάδελφος ο κύριος Σούκορ με αντικατέστησε. Δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι παρόν. Λυπάμαι γι' αυτό. Τώρα αν μου να κάνω μία σύνοψη της κατάστασης. Έλαβα 68 τροπολογίες. Μεγάλος αριθμός. Εξεπλάγει να πω την αλήθεια. Από 7 συναδέλφους. Και εγώ ίδιος ε, είμαι νομικός. Και να πω ότι στατιστική δεν είναι, αν θέλετε, και το θέμα το οποίο είμαι Όμως τώρα, μετά τη μελέτη που έκανα, έχω μια καλύτερη εικόνα για το ζήτημα αυτό. 12 τροπολογίες έρχονται να τροποποιήσουν τις δικές μου τροπολογίες. Ουσιαστικά είναι 56 ουσιαστικά νέες τροπολογίες για νέες προσθήκες ή αλλαγές. Θα πω ευθύς εξ αρχής ότι συμφωνώ σχεδόν με όλες ε, αυτές τις τροπολογίες απόλυτα. Γιατί οι τροπολογίες αυτές συμβάλλουν στην αύξηση αποτελεσματικότητας των στατιστικών δεδομένων και καθεστούν σαφές, σαφώς συγγνώμη, τι, ποιους δείκτες χρειαζόμαστε για να μπορούμε να συλλέγουμε καλύτερα συστικά στοιχεία. Να σας πω τώρα, χθες έλαβα και ε, την γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το, για το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Οι σκιώδες δεν έχουν λάβει ακόμη αυτό το κείμενο της Κομισιόν, έτσι νομίζω θα τους το διαβάσω πάντως. Από αυτό το κείμενο, την επιστολή ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ εξήγα το συμπέρασμα ότι ε, η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρνητική έναντι της γνωμοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολείπεται σημαντικά ως προς τη μέθοδο συλλογής δεδομένων. Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό και την καταπολέμηση της φτώχειας και εκεί βλέπουμε καθυστερήσεις. Το 2014-2015 θα είναι έτοιμη η Κομισιόν. Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, τροπολογίες, συμφωνώ με τις τροπολογίες εκείνες που αφορούν την αποτελεσματική χρήση των δαπανών, με την αποτελεσματικότητα εν γέννη, με τις διαδικασίε πιστοποίησης. Ε, υπάρχουν 9-10 τροπολογίες που αφορούν τη συλλογή δεδομένων ε, για θέματα πέρα από την απασχόληση. Έπειτα υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που έχουν ως αντικείμενο τη μείωση των δαπανών, χωρίς όμως να είναι πολύ συγκεκριμένη πρόταση που κάνουν. Θεωρώ, λοιπόν, ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό, σε συμβιβαστικά τροπολογίε που έχουν στόχο την αποτελεσματικότητα τη χρήση των δαπανών και εκεί θα υπάρχει συμφωνία, ελπίζω. Συνολικά λοιπόν από τις 68 τροπολογίε, 7 ίσως είναι προβληματικές. Για τις υπόλοιπες είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις ή να υποστηρίξουμε ε, απόλυτα αυτές τις τροπολογίες και έτσι να υποστηρίξουμε την γνωμοδότηση. Από κοινού τους οικειώδεις συζητητές παρακαλώ να υποστηρίξετε αυτή τη γνωμοδότηση αλλά θέλω και τη δική σας συμβολή με τις δικές τοποθετήσεις για να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω σημειώσει την κυρία Παπαδοπούλου που έχει ζητήσει το λόγο. Thank you very much. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια από, τις, από την ομάδα των σοσιαλιστών. Πρώτα, συγχαίρω τον κύριο Κώσα για τη έκθεση του. Συμφωνεί με πολλές από τις δικές μας τροπολογίες. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα είναι το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις δραστηριότητες της Ευρωστάτ, όπως προβλέπεται και στην πρόταση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που εκρήθηκε τον Ιούνιο. Δεν έχουμε λάβει ακόμα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το γεγονό ότι ο κ. Κώσα, το είπε άλλωστε προηγουμένως, ότι αυτό είναι αρνητικό, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους και οδησίγητες αλλά και ανυπομονησία να λάβουμε στα χέρια μας την γνωμοδότηση αυτή το δυνατόν συντομότερο. Θέλουμε να δούμε δηλαδή ποια είναι η άποψη τη Κομισιόν. Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι το θέμα δεν είναι επίμαχο. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα να δούμε ποιου συμβιβασμού προτείνει ο κ. Κώσα. Και είναι απαραίτητο να διεξαχθεί το δυνατόν συντομότερο συνάντηση για να ακούσουμε τις απόψεις του για τις 68 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από όλες τις πολιτικές ομάδες. Προσωπικά έχω εγώ καταθέσει 19 τροπολογίες από, ε, για λογαριασμό της ομάδας μου δηλαδή που ελπίζω ότι δεν θα ε, αποτελέσουν πρόβλημα και σε αυτές τονίζουμε την ανάγκη να είναι υψηλής ποιότητας τα στατιστικά δεδομένα σε όλους τους κέριους τομείς για την καινοτομία και την ανανέωση, για την ενέργεια, τις μεταφορές, το περιβάλλον και όλους τους άλλους κέριους τομείς των κοινωνικών πολιτικών. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα θα παραμείνει πάροχος υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στατιστικής. Χρειαζόμαστε βέβαια ενιαίες προδιαγραφές, ενιαία πρότυπα που να βασίζονται στην ε, προσβασιμότητα, στην συνοχή και βεβαίως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές θα εξυπηρετούν τα ενδιαφέροντα όλων των χρηστών, βεβαίως αυτών που ασκούν την πολιτική, των ερευνητών, των επιχειρηματιών, των αρχών και ούτω καθεξής. Και επομένως οι ευρωπαϊκές στατιστικές δεν θα είναι μοναχά υψηλής ποιότητας, αλλά και προσιτές σε όλους. Εν τέλει, μία από τις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς είναι ότι το δημοσιονομικό δελτίο του προγράμματος θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύπτει τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των διαδικασιών, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας στατιστικών δεδομένων και στο εθνικό επίπεδο, αλλά και για την εκπαίδευση των εθνικών στατιστικολόγων. Αυτό είναι λίγο πολύ το νόημα των τροπολογιών που έχουμε καταθέσει και αναμένουμε βεβαίως με ενδιαφέρον τη συνάντηση μεταξύ εισηγητού και σχεδόν εισηγητών όπου θα διεξαχθεί συζήτηση για να δούμε πώς προτίθεται να προχωρήσει με τις συμβαστικές τροπολογίες. Και βέβαια θα χρειαστούμε, όπως είπα και πριν, το δυνατόν συντομότερο την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Μπένιανε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον εισηγητή και τους συναδέλφους του για το έργο τους και για αυτές τις τροπολογίες. Οι περισσότερες τροπολογίες ε, θα έχουν την υποστήριξή μου και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες ε, κάπου στη μέση που θα ήταν καλύτερα για συμβιβαστική τροπολογία. Ορισμένες ωστόσο τροπολογίες ε, που προκαλούν επιφυλάξεις. Οι 19 και 21 όπου γίνεται έκκληση για μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Πιστεύω είναι σημαντικό η συλλογή δεδομένων και οι κοινωνικοί δείκτες ε, που έχουν ήδη ληφθεί υπόψη σε στατιστικά προγράμματα από τα κράτη-μέλη έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τα κράτη-μέλη και ουσιαστικά προσπαθούμε να τους πούμε πού πρέπει να εστιάσουν το έργο τους. Αυτό είναι δύσκολο πιστεύω. Η στατιστική μέθοδος δηλαδή που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει λοιπόν να αποφασιστεί πώς θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αφού συλλεχθούν. Δεν χρειάζεται να λέμε να, στους ε, υπευθύνου συλλογή δεδομένων. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να διατηρήσουμε ως αρχή με ανήσυχη η πολιτικοποίηση της συλλογή δεδομένων. Μπορούμε να είμαστε όσο πολιτικοί θέλουμε αφού τα συλλέξουμε και αφού τα αναλύσουμε. Ωστόσο η συλλογή δεδομένων και η ανάλυση ίδια θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από πολιτικές απόψεις. Θα πρέπει να είναι αντικειμενικές. Αυτό ισχύει επίσης για τις τροπολογίες 53, 54, 60 και 61. Δεν θέλω να θέσω σε κίνδυνο την αντικειμενικότητα της Eurostat φέρνοντας πολιτικά στοιχεία. Η τροπολογία 22 πιστεύω είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες όταν δημιουργούμε επιπλέον απαιτήσει. Υποστηρίζω λοιπόν την Κομισιόν που προσπαθεί να μειώσει τη γραφειοκρατία. Προτιμώ λοιπόν το αρχικό κείμενο από την τροπολογία. Όσον αφορά την τροπολογία 23, δεν υπάρχει κάτι κακό στο να ανοίξουμε τα προγράμματα στις ε, χώρες του 7. Φυσικά δεν μπορούμε να τους το επιβάλλουμε εφόσον χρησιμοποιούν παρόμοιες μεθόδους ε, ώστε να μπορεί να γίνεται σύγκριση και θέλουν να συμμετέχουν, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Δεν υποστηρίζω λοιπόν την 23. Δεν κατάλαβα την ε, τροπολογία 25 για το παράρτημα. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για, το, για ποιο λόγο θα απαιτείται κάτι τέτοιο. Στην τροπολογία 56 Πιστεύω ότι οι κοινωνικές ανησυχίες ε, πιστεύω ότι η τροπολογία αυτή δεν είναι κατάλληλη. Δεν υποστηρίζω την 56, δηλαδή η 69 και 71. Εκεί αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε παραδείγματα με τους Ρωμάς του 69 Πιστεύω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε παραδείγματα, διότι υπάρχουν πολλές μειοψηφίε και πολλές κατηγορίες και χρησιμοποιώντας παραδείγματα αρχίζουμε να δημιουργούμε λίστες ανθρώπων και κάποιοι θέλουν να ξέρουν γιατί αυτοί δεν έχουν συμπεριληφθεί στην λίστα ενώ άλλοι έχουν συμπεριληφθεί. Συνεπώς δεν ε, υποστηρίζω αυτές τις τροπολογίες για αυτούς τους απλούς λόγους. Παρότι θα ήθελα να συμπεριληφθούν οι Ρωμα φυσικά στις μειονότητες καθώς και οι χαμηλά αμοιβόμενοι εργαζομένοι στις κατηγορίες. Αυτή είναι η τελευταία παρατήρηση μου. Ευχαριστώ. So, vielen Dank. Jetzt, ähm, Ευχαριστώ λοιπόν. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κανείς παρόν. Το όνομα που μου έχουν δώσει είναι του κυρίου Γιώχαμ Ρέχτενβαλτ. Έχετε το λόγο, αγαπητή κυρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελε να ευχαριστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εισηγητή κ. Κώσα, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης για το έργο που έχουν επιτελέσει επί του σχεδίου κανονισμού και όπως τόνισε ο εισηγητής σας και το τόνισαν και οι σκιώδεις εισηγητές που μίλησαν, είναι σημαντικό το νομοθέτημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία διότι προσφέρει την βάση για την εργασία τα επόμενα χρόνια. Έχει σχεδιαστεί με τρόπο που αποδίδει η σημασία στις ανάγκες στατιστικών δεδομένων για τους τομείς απασχόλησης και κοινωνικών πολιτικών και από την άλλη μεριά για τις οικονομικές πολιτικές. Υποτίθεται δηλαδή ότι θα είναι ισότιμες οι στατιστικές αυτές. Η σημασία του νομοθετήματος υπογραμμίζεται και από τον αριθμό και την φύση των τροπολογιών που έχουν καταθέσει τα μέλη της Επιτροπής σας. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να συμφωνήσει με μεγάλο αριθμό των τροπολογιών αυτών, ωστόσο για ορισμένες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτιμήσει να διατηρήσει την αρχική διατύπωση και, ή θα προτείνει συμβαστικές διατυπώσεις λαμβάνοντας υπόψη ε, διάφορες τροπολογίε για το ίδιο θέμα. Διαρωτώ λοιπόν κυρία Πρόεδρε εάν υπάρχει δυνατότητα να σας δώσει η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή στα μέλη της Επιτροπής σας τις επόμενες ημέρες πιο λεπτομερείς αντιδράσεις της για τα θέματα όπου ε, διστάζει ακόμα να συμφωνήσει. Όπως ακούσατε, το περιμένουμε αυτό εδώ και καιρό, λέει η Προεδρεύουσα κυρία Σρέντερ. Τώρα, ο κύριος Κώσα παρακαλείται να συνοψίσει και ενδεχομένως να απαντήσει στο α ή β θέμα εφόσον το επιθυμεί. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την τοποθέτησή τους και σε ό,τι μια φορά θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστείλει σε εμένα και σε όλους τους κοιόδης όλα τα σχόλια και παρατηρήσεις της, διότι πρέπει να κλείσει σύντομα οποιαδήποτε διεργασία για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης γιατί θα κλείσει ο φάκελος. Ε, σε ό,τι με αφορά, συμφωνώ με τους δύο σκιώδεις, επιβεβαιώνω και εγώ τα λεγόμενά τους και εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία τροπολογιών δεν είναι προβληματικές. πρέπει θα πρέπει να έχουμε παρακολούθηση καλύτερης ποιότητας και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη διαδικασία εχνηλάτησης του κόστους. ώστε να μπορούν να καλύπτεται πλήρω οι δαπάνες. Άκουσα και κάποιες επιφυλάξει για κάποιε τροπολογίε. και εγώ συμφώνω. Δεν είπα ότι διαφωνώ κάθετα με κάποιε τροπολογίε. Πιστεύω ότι μπορούμε σε μία συνάντηση στο άμεσο μέλλον με τους κοιόδες ηγητές θα μπορέσουμε να βρούμε μία ε, καλή λύση για αυτά τα ζητήματα που δημιουργούν δισταγμούς. Μιλάμε για πέντε εξτροπολογίες ε, ουσιαστικά τις οποίες εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω. Γιατί ο βασικός ο στόχος είναι να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Ε, οπότε δεν έχω σοβαρά προβλήματα για κάτι τελευταίο. Η επιστολή που έλαβα χθε δεν είναι αρνητική ε, γνώμη της Κομισιόν, το συμπέρασμα που έβγαλα από αυτή την επιστολή είναι το εξής. Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και σε ό,τι αφορά τον αγώνα για την ε, κοινωνική ένταξη, η Eurostat υπολείπεται. Ε, είναι ο αρμόδιος οργανισμός και συλλογή δεδομένων η Eurostat ούτως ή άλλως. Και θεωρώ ότι η Επιτροπή Απασχόλησης έχει ως ε, βασικό σκοπό να δραστηριοποιηθεί σε αυτούς τους τομείς και για να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε χρειαζόμαστε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Επίσης, είμαι της γνώμης ότι τέτοιου είδους καθυστερήσεις ε, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές ε, στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά αυτό το, μάλλον τους συμβαστικές μου προτάσεις τις αποστείλω το στομότερο δυνατόν στους σκιώδεις και πιστεύω και τα λοιπά θα μπορέσουμε να βρούμε σίγουρα μια λύση. Θα σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας και προσβλέπω στο περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μήνα χρόνο διαθέτεται για να κάνετε τη σχετική διαπραγμάτευση. Τέλη Μαΐου θα πρέπει να έχουμε φτάσει σε επίπεδο που να μπορούν να υποβληθούν οι ε, συμβασικές τροπολογίες, να γίνει η ψηφοφορία στις 31 Μαΐου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις προσπάθειες. Και αυτό ήταν βεβαίως το τελευταίο μας θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ευχαριστώ όλες και όλους που μείνατε μέχρι τέλους της συνεδριάσεως εδώ. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Θα συνεδριάσουμε ξανά 30 και 31 Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ.